il Καλή σα ημέρα κυρίε και κύριοι, αρχή της συνεδρίασης. Βάσει της ημερησία διατάξεως, πρώτο σημείο έχουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Θα δώσω αμέσως το λόγο ε, στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου, στην Υπουργό κυρία Μπερντιάκ Νικολίνα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Και βεβαίως ε, θα ήθελα ε, να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία της την κυρία Σουίτσα, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίες, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία ε, να συζητήσουμε για το θέμα της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως σας είπε και ο Πρωθυπουργό χθε, ε, όσον αφορά το Συμβούλιο, ξεκινούμε να εργαζόμαστε ε, έτσι ώστε να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες για την διάσκεψη. Ξέρετε ότι ήδη από τον Δεκέμβριο υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το θέμα αυτό. Προτεραιότητα ότι θα δοθεί στην υλοποίηση της στρατηγικής ε, ε, ατζέντα ε, για την επόμενη περίοδο. Και βεβαίως θέλουμε να εργαστούμε για το καλό των πολιτών. Οι προτεραιότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στη στρατηγική ατζέντα απηχούν τους προβληματισμούς των πολιτών. Η διάσκεψη θα πρέπει να βασιστεί και στους διαλόγους που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, και βεβαίω ε, ήδη έχει υπογραμμιστεί ο τρόπο με τον οποίο η διάσκεψη αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να στεφθεί από επιτυχία έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να δούμε τι στρατηγικέ μας μέσω και μακροπρόθεσμα και να αντιμετωπίσουμε έτσι τις προκλήσεις της Ευρώπης. Οπωσδήποτε η διαδικασία δε που θα οδηγήσει στην, στην διάσκεψη θα πρέπει να είναι συμπεριληπτική έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα κράτη-μέλη με ίδιο τρόπο συμπεριλαμβανομένων δε και των κοινοβουλίων τους αξιότιμοι βουλευτές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Κροατική Προεδρία ε, να εργαστεί ε, για την θέσπιση κοινή ε, θέσης όσον αφορά την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και να εμπλακεί με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί τη βάση αυτών. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την εργασία και μπορώ να σας πω ότι ήδη σήμερα στις Βρυξέλλες οι πρέσβεις έχουν την πρώτη ανεπίσημη εντελεγή απόψεων για το θέμα αυτό. Στην, ε, ε, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 28ης του μηνός θα συζητηθεί το θέμα ε, και βεβαίως προσδοκώ να παρακολουθήσω τις συζητήσεις σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα παρακολουθήσω τα λεγόμενά σας με προσοχή έτσι ώστε να δώσω και το απαραίτητο input στη διάσκεψη της επόμενης εβδομάδας. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος και τώρα θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο κυρία Σουίτσα. Παρακαλώ κύριε Σουίτσα, έχετε το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί Υφυπουργέ, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ε, με τιμά το, ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας για να συζητήσουμε το μέλλον της Ευρώπης και ως πρώην Ευρωβουλευτής θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας πολύ στενός φίλος και βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας και πάλι ως φίλος αλλά και ως ε, εταίρος ε, ε, με βάση τη νέα μου ιδιότητα της Επιτρόπου Αρμόδιας για θέματα δημοκρατίας και δημογραφίας. Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για τους πολίτες η Ευρωπαϊκή Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία, γιατί στη τελική ανάλυση για το δικό του συμφέρον λαμβάνουμε αποφάσεις. Αν και μερικές φορές κάνουμε και λάθη και θα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Τώρα όμως έχουμε την ευκαιρία να αφουγκραστούμε τους πολίτες, να ακούσουμε τη γνώμη τους, να δώσουμε απαντήσεις, εξηγήσεις, διευκρινήσεις, να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα δούμε περί τίνος πρόκειται όταν μιλούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε σε κρίσιμη ιστορική στιγμή της ευρωπαϊκής ιστορίας και έχουμε μια μοναδική ευκαιρία και πολλές προκλήσεις. Και αν τα καταφέρουμε, οι συνέπειες θα επηρεάσουν όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον. Οπότε αναπόκειται σε όλους μας ε, να εργαστούμε ώστε να στεφθεί με επιτυχία αυτή η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Και ας είμαστε σαφείς, ε, ο παλιός τρόπος άσκησης πολιτικής δεν λειτουργεί πια. Δεν είναι τύχες για τυχα πάντα. Θα πρέπει να ακούσουμε τους πολίτες, ε, να τους δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται. Συνεργασία και κουράγιο είναι οι λέξεις κλειδιά της νέας διαδικασίας. Θα πρέπει να είμαστε γενναίοι και να βρούμε νέες δημιουργικές ευρηματικές λύσεις για να λειτουργήσει η δημοκρατία μας ακόμη καλύτερα για τους πολίτες. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε από κοινού, ως εταίροι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό μια κοινή διακήρυξη και των τριών θεσμικών οργάνων μπορεί να χαράξει το δρόμο για αυτή τη μοναδική εταιρική σχέση Βέβαια, μια εταιρική σχέση δεν σταματά στα τρία θεσμικά όργανα. Τα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει επίση να αναμειχθούν στη διαδικασία αυτή. Η συνεργασία του θα είναι ένα του αυτή τη διαδικασία. Και για να είμαστε σίγουροι ότι θα αγγίξουμε όλου του πολίτε, ε, ακόμη και αυτούς που δεν έχουν άμεση επαφή μαζί μα. Ε, θα στηριχθούμε στη συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Μάλιστα, ω Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα επισκεφτώ και τι περιφέρειε. Θέλω να ακούσω του πολίτε από την κάθε γωνιά τη Ευρώπη. Και θα σταματήσουμε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Όχι, βέβαια, πρόκειται για μια ανοιχτή διαδικασία. Και όσο προχωρά η διάσκεψη, φαντάζομαι και άλλοι θα λάβουν μέρο. Και έχουμε δύο άξονε στη συζήτηση. Μία συζήτηση πολιτική γύρω από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το στρατηγικό θεματολόγιο του Συμβουλίου και ο δεύτερος άξονας αφορά θεσμικά ζητήματα όπως την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια. Εδώ ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι ο ρόλος ενός έντιμου διαμεσολαβητή και η Βέρα Γιούροβα, η συνάδελφος επίτροπος, θα παρακολουθήσει αυτό το θεσμικό άξονα της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει τη δική της πρόταση στις 30 ε, Ιανουαρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Και αυτή θα είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στις συζητήσεις που θα γίνουν στις επόμενες εβδομάδες μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να συμφωνήσουμε από κοινού για το πεδίο εφαρμογής, τη μορφή, τη δομή και το στόχο της διάσκεψης. Και αυτό θα είναι το περιεχόμενο της κοινή διακήρυξης που σας προανέφερα. Και ενώ το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα συζητήσει ε, στις 28 Ιανουαρίου τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, εμείς θα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη δεύτερη φάση και να προσδιορίσουμε την ημερομηνία έναρξης της διάσκεψης, ε, ελπίζουμε κατά το πρώτο εξάμεινο του 2020. Και η καλύτερη νομίζω ιδεώδης ημερομηνία για την έναρξη θα ήταν η 9η Μαΐου, η μαιου η μέρα της Ευρώπης. Μία πολύ συμβολική και σημαντική για μας μέρα. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό για μια καρποφόρα συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έχουμε πολλές κοινέ προτεραιότητες. Και εγώ ως αντιπρόεδρος, ε, μάλιστα ο Μάρος Σεφτσοβιτς ως αντιπρόεδρος ε, αρμόδιος για τις διακοινοβουλευτικές ε, σχέσεις, επίση θα λάβει μέρο στη συζήτηση. Και εσεί, ω άμεσα αιρετή εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, θα έχετε κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Και χαιρετίζω το ψήφισμά σα, αλλά και τη δέσμευσή σα να μην προεξοφλήσουμε την έκβαση της διάσκεψης το, κάτι τέτοιο, προδικάσουμε το, το αποτέλεσμα της α, διάσκεψης θα είναι πολύ αρνητικό για τη δημοκρατία. Είναι πολύ χειρότερο από το να μην κάνουμε απολύτω τίποτα. Δεν θα προεξοφλήσουμε τίποτα λοιπόν. Και με την επιβεβαίωση ε, του διορισμού μου, μου δείξατε εμπιστοσύνη. Και είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη και στους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά θέλω να κερδίσω και τη δική σας εμπιστοσύνη και στο μέλλον. Γι' αυτό και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Και πριν δώσω τον λόγο εις τους Προέδρου των πολιτικών ομάδων θα ήθελα να πω δύο λόγια. Εδώ και μήνε εργαζόμαστε ε, για αυτό το θέμα της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και βεβαίω, είμαι ιδιαίτερο ευτυχή, ε, που σήμερα ε, διεξάγεται αυτή η συζήτηση ε, στα, και ε, το γεγονός ότι ε, θα ψηφίσουμε αργότερα και το ψήφισμα για την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Γνωρίζετε ότι προέκυψε η διάσκεψη αυτή μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάγεν, ε, ε, θεώρησε ότι ε, έπρεπε να την συμπεριλάβει το πρόγραμμα. Υπάρχουν μηχανισμοί της ευρωπαϊκής δημοκρατικής διακυβέρνησης. Έχουμε διαπιστώσει ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν, να μεταρρυθμιστούν και θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα Εθνικά Κοινοβούλια και σε μια διαδικασία ακρόασης των ε, προβληματισμών των πολιτών. Ε, θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα ξεκινήσει μία διαδικασία μεταρρύθμισης που δεν θα έχει προδικαστεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ε, χρειαζόμαστε ε, μια λειτουργική δημοκρατία, μια δημοκρατία που θα λειτουργεί σωστά. Χρειαζόμαστε μια δημοκρατία η οποία θα βαίνει προς όφελος των πολιτών. Πιστεύω ότι αυτό είναι και προς όφελος ε, των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν τέλει προς όφελος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς εμείς ανοίξαμε το δρόμο στους πολίτες και πιστεύω ότι σήμερα είναι πολύ σημαντικό σημαντική ημέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί μαζί με όλες τις πολιτικές ε, ομάδες ξεκινούμε αυτήν την διαδικασία, αυτήν την διαδρομή διαλόγου ε, μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επιτύχουμε εάν και εφόσον όλα τα θεσμικά όργανα ακολουθήσουν αυτήν την κοινή πορεία. Ε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον κύριο Μάνφρετ Βέμπερ, πρόεδρο του ΕΛΚ. Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, εκπρόσωποι του Συμβουλίου, το σημείο εκκίνηση για τη συζήτησή μα για τη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών ε, πέρσι. 201 εκατομμύρια πολίτε ήρθαν στι κάλπε. Η δεύτερη μεγαλύτερη δημοκρατία στη γη. Αυτό ήταν το σημείο εκκίνηση, λοιπόν. Οι άνθρωποι πιστεύουν και πιστεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να διαμορφώσουν το μέλλον τη. Το βασικό λοιπόν ερώτημα τώρα είναι κατά πόσον μετράει η ψήφο μου. Αλλά κατά πόσον έχει αντίκτυπο. Και εδώ ξέρουμε ότι ε, επιτέχεται βελτιώσεων το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να είναι μια δεκαετία ενίσχυσης της ε, ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ποιε είναι οι αρχές για την ε, εργασία μας ως ΕΛΚ. Το πρώτο και βασικό σημείο, όπως αναφέρθηκε, είναι η συμμετοχή του κόσμου. Να βρούμε έναν τρόπο να αγγίξουμε τις ιδέες και τις αντιλήψεις του κόσμου, του εκλογικού κοινού. Κατά δεύτερον, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ε, στην πρώτη θέση. Εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι των πολιτών, εμείς εκπροσωπούμε το πολιτικό τοπίο πολιτικά και γεωγραφικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπροσωπούμε ένα κοινοβούλιο όπου πραγματικά σεβόμαστε την ελεύθερη εντολή και είναι δύσκολο για μένα ως επικεφαλής της ομάδας μου να πετύχω ε, ομοφωνία στην ομάδα μου. Είναι καλό αυτό γιατί πραγματικά εκπροσωπούνται όλα και επίσης ε, καλές σχέσεις ε, εργασίας με το Συμβούλιο. Η κυρία Ντουμπράφκα μπορεί πραγματικά να συνεργαστεί μαζί μας, να υπολογίζει τη συνεργασία αυτή μαζί μας. Και ένα άλλο στοιχείο είναι να συμμετέχουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όλα αυτά είναι συμπεριφωνημένα, αλλά και πάλι θέλουμε να πούμε ότι η διαδικασία διαμόρφωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των κοινοβουλίων είναι για μα το κλειδί. Ύστερα το θέμα τη κατεύθυνση. Η δημοκρατία βασίζεται σε δύο αρχέ, στου υποψηφίου και στο πρόγραμμά του. Θα πρέπει να δούμε ότι αυτό ισχύει για τους δημάρχους, για τους καγκελάριους, αλλά και για μας. Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, σε ό,τι αφορά τη θέση της Πρόεδρου και του Πρόεδρου α, της Επιτροπής. Και η διαδικασία του επικεφαλής υποψηφίου, του Σπίτσεν Καντιντάτα, πέρσι απέτυχε, αλλά θέλουμε ε, ως ΕΛΚ να καταστεί η διαδικασία αυτή δεσμευτική για τις επόμενες εκλογές. Χρειάζεται ε, υγιή συνταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, πολιτικών ομάδων. Θα πρέπει να αντικαταπτρίζονται λοιπόν και οι κανόνε για τα πολιτικά αυτά κόμματα, για τα ε, πολιτικέ ομάδε. Και θα πρέπει να δούμε πώ θα ενισχύσουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου το δικαίωμα, για παράδειγμα, τη πρωτοβουλία. Θα πρέπει να το κατοχυρώσουμε καλύτερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω και για τα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια. Πιο πολύ δημοκρατία, λοιπόν, και να αποφασίζει ο κόσμο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο κατά τη τάση των αντιευρωπαϊστών. Και τέλο, είμαστε προετοιμασμένοι για τις ε, προκλήσεις του αύριο, πραγματικά προετοιμασμένοι. Τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της Τρεχούσα συνθήκη και επίσης χρειάζεται ε, αλλαγή των συνθήκων. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα για το μέλλον της Ευρώπης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα, ας συνεργαστούμε για να έχουμε ένα καινούργιο όραμα και όνειρο για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η πρόεδρος ε, ε, Γκαρθία Πέρες, από ε, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κύριε Πρόεδρε, στις 9 Μαΐου θα έχουν περάσει 30 χρόνια από τη διακήρυξη του Σούμαν και τότε ξεκινούσε μια πολιτική διαδικασία στην ιστορία και σε όλο τον κόσμο οι ε, ορισμένες χώρες αποφάσισαν ε, να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών τους ε, και να πορευτούν μαζί. Και βεβαίως η Ευρώπη δεν οικοδομήθηκε σε μία μέρα, αλλά σε μία διαδικασία επί τη βάση της αλληλεγγύης. Εμείς τώρα πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση σε αυτήν την Ευρώπη, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών και να επικρατήσει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα όπως είναι η ψηφιοποίηση, η κλιματική αλλαγή κλπ. Ε, αλλά υπάρχουν και ε, λαϊκιστικές επιθέσεις ε, οι οποίες αλλοιώνουν τις διαδικασίες. Δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε, να αποστρέψουμε το βλέμμα από αυτές τις προκλήσεις. Πρέπει να δώσουμε βέβαια και μια ευκαιρία στους πολίτες να μιλήσουν, να ακούσουμε τις προσδοκίες τους, να ακούσουμε τις προτάσεις ε, που έχουν να υποβάλουν, να ακούσουμε όλα τα πεδία της ε, κοινωνίας, όλους τους τομείς της κοινωνίας. Ε, άλλωστε αυτή ήταν και η μεγάλη αρχή της διάκρισης της Χάγης του 1948 ε, και θα πρέπει να δώσουμε ε, και ε, τον λόγο στην κοινωνία των πολιτών. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες θέλουμε να προκύψει ένας πραγματικός διάλογος με την κοινωνία από τον οποίο θα απορρεύσουν συγκεκριμένες προτάσεις και αυτή η συζήτηση να γίνει σε πλήρη ισορροπία γεωγραφικής προέλευσης ε, ε, ε, οποιασδήποτε άλλης προέλευσης η ισορροπία των φύλων κλπ. Δεν υπάρχουν πρώτες ή δεύτερες κατηγορίες πολίτες ή χώρες ή πόλεις. Εμείς, όπως έλεγε και ο Ζαμονέ, δεν είμαστε εδώ για να χωρίσουμε τον κόσμο και να τον αξιολογήσουμε, αλλά για να ενώσουμε τον κόσμο. Ε, θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια Ευρώπη η οποία ενωμένη θα μετρήσει περισσότερο γιατί έχει μεγαλύτερο βάρος μια ενωμένη Ευρώπη και αυτό θέλουμε. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε ε, την ε, Ευρώπη και δεν θέλουμε εμείς εδώ να οικοδομήσουμε ή να ενδυναμώσουμε μια αγορά. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Για, δυστυχώς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέστρεψε το βλέμμα από αυτές τις ε, ε, διαδικασίες. Ε, άφησε να μεγαλώσει και η φτώχεια και οι ανισορροπίες και άφησε χώρο για να αναπτυχθεί ο λαϊκισμός. Πρέπει να δώσουμε μια όθηση λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη συνθήκη της Λισαβόνας που ήδη ενδυνάμωσε τις διαδικασίες, ωστόσο δεν ήρκεσε. Ε, ελπίζουμε ότι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ε, θα ανοίξει νέα πεδία εμπλουτισμού της κοινωνίας ε, και άλλα στοιχεία τα οποία θα βελτιώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές του 2024. Ε, έχουμε πορευτεί σε μια πολύ μεγάλη πορεία. Έχουμε διευρύνει την ευρωπαϊκή οικογένεια. Ε, καταφέραμε να είμαστε 28. Δυστυχώ. θα αποχαιρετήσουμε με μεγάλη θλίψη ε, μια χώρα και αυτή είναι μια καλή χρονική στιγμή, μια καλή ευκαιρία για να ξανασυζητήσουμε τις διαδικασίες και τη βάση της Ευρώπης. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε αυτά που μας ενώνουν, αλλά πρέπει να έχουμε και συνείδηση ότι εμείς κρατάμε στα χέρια μας το μέλλον. Όχι, δεν χρειάζεται να ε, πέσουμε στην, ε, σε μια νοσταλγική αναπόλυση του παρελθόντος της Ευρώπης. Το μέλλον μας ανήκει και εμείς ε, όλες και όλοι θα πρέπει να καθορίσουμε το μέλλον. Εμείς σαν σοσιαλιστές και δημοκράτες θα βάλουμε το λιθάρι μας για να οικοδομηθεί αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος Τσιόλος για την ομάδα Renew Europe. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Πολύ συχνά λέμε εδώ ότι η πολυμορφία είναι ένα του της Ευρώπης. Ε, τώρα έχουμε την ευκαιρία να το αποδείξουμε κιόλα. Οι ευρωεκλογέ έχουν δείξει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε πιστεύουν στην Ευρώπη. Θέλουν όμω μια καλύτερη ε, Ευρώπη και ανανεωμένη. Οπότε η πρώτη αλλαγή θα πρέπει ε, να είναι στον τρόπο που θα εμπλέξουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί η Ευρώπη δεν έγινε για μια ελίτ, για τις Βρυξέλλες, για μια ομάδα, αλλά για να υπηρετήσει όλους τους πολίτες. Οπότε η διάσκεψη μπορεί να γίνει μια καταπληκτική ευκαιρία ανανέωσης της Ευρώπης και αναζωογόνησής της. Αν ε, έχουμε το κουράγιο να ξεφύγουμε από το διαδικαστικό μας τρόπο σκέψης και να δώσουμε το λόγο στους πολίτες. Για πολλά χρόνια αφήσαμε να αναπτυχθεί συχνά ένα αίσθημα ότι η Ευρώπη κοφεύει ότι επιβάλλει κανόνες και περιορισμούς. Και η Ευρώπη που οικοδομεί είναι κρυμμένη πίσω από μια Ευρώπη περιορισμών. Η διάσκεψη θα είναι μια ευκαιρία για να ανοίξουμε διάπλατα τις πόρτες της Ευρώπης προς τους πολίτες. Και δεν είναι τυχαίο που είμαστε υπέρ της ημερομηνια 9 η Μαΐου για την έναρξη αυτής της διάσκεψης. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις για να εμπλέκουμε τακτικά τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι μία φορά κάθε πενταετία για τις ευρωεκλογές. Βέβαια κάποιοι ανησυχούν γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν κάποιες ε, ευθύνες και αρμοδιότητες. Όμως ε, είμαι πεπισμένος ότι η συμμετοχική δημοκρατία και η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι συμπληρωματικές έννοιες και όχι αντικρουόμενες. Έχουμε δυόμιση χρόνια για να καταθέσουμε ιδέες και προτάσεις που θα καταστήσουν όχι μόνο πιο αποτελεσματική τη λειτουργία των θεσμικών μας οργάνων και πιο εύληπτη, αλλά θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όσων θέλουν να γίνει ένας πραγματικός κοινό σήκος η Ευρώπη. Γιατί πολλοί ε, αρχίζουν και αδιαφορούν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα συνδυάσουμε το σύνδεσμο με μια συγκεκριμένη κουλτούρα, με ένα συγκεκριμένο χώρο και περιοχή, με την ευρωπαϊκή ταυτότητα, γιατί είναι και τα δύο ταυτόχρονα Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 10 χρόνια από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και ταυτόχρονα έχουμε και το Brexit. Δεν θα ήθελα να το συνδέσω, αλλά ήρθε η ώρα να αναζωογονήσουμε την Ευρώπη και να την προσαρμόσουμε στις προκλήσεις του σήμερα. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε το σύνδρομο της ευρωπαϊκής φούσκας, της ευρωπαϊκής Οφόλικα. Θα πρέπει να προωθήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το νέο όραμα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο ε, στον ε, κύριο Φρόιντ των Πρασίνων και μετά Τζάνι για την ταυτότητα και δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση που έχουμε σήμερα είναι ε, ένα δώρο για τον Άιτζελ Φαράζ. Γιατί τι καλύτερο για την τελευταία ολομέλεια να αφιερώσουμε μεγάλο χρόνο στη συζήτηση στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης που είναι ο χειρότερος του εφιάλτης. Κρίμα λοιπόν που δεν είναι παρόν. Γιατί μας αποκάλεσε φεδεραλιστική κλίκα και φεδεραλιστική συνωμοσία. Κι όμως ε, είναι μια δημόσια δημοκρατική διαδικασία, όχι ε, μια παλιά ιδεολογία. Γιατί η αλληλεγγύη είναι ισχυρότερη από το μίσο και η συνεργασία είναι ισχυρότερη από τον εθνικισμό. Και όταν ε, ο Νάιτζελ και η κλίκα των, ψευτο, των ψευτών υπέρμαχων του Brexit ε, οδήγησαν την, ε, την ε, Μεγάλη Βρετανία έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέλουμε μια ισχυρότερη δημοκρατική ένωση γιατί έχουμε πολλές ανισότητες, αδικίες, τις μεγάλες εταιρείε να μην πληρώνουν τους φόρους τους, μια, μια Αμερική που απομακρύνεται, μια Κίνα που αυξάνει την επιρροή της. Δεν είναι ώρα για εθνικούς εγωισμούς. Θα πρέπει να ενωθούμε, θα πρέπει να συνεργαστούμε Ιδεμή θα χαθούμε μόνοι και απομονωμένοι. Γι' αυτό οι προτάσει που καταθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ισχυρέ, Στηρίζονται στα καλά παραδείγματα που είδαμε στην Ιρλανδία, ε, στι ε, συνελεύσεις των πολιτών και φιλοδοξούμε να έχουμε ευρία συζήτηση με τους πολίτες από όλη την Ευρώπη, με τα εθνικά κοινοβούλια, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και τους συντηρητικούς ότι δεν αρκεί να έχουμε την Business Europe και τους κοινωνικούς εταίρους για τα συνδικάτα στις συζητήσεις. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις στη συζήτηση. Και γνωρίζω ότι ελοχεύουν κίνδυνοι στη διαδικασία, γιατί θα έχω μια συζήτηση σε 24 γλώσσες. Ίσως μπορεί να μην ε, σπάσουμε μέσω στη φούσκα των Βρυξελών και να, ε, να προτείνουμε τις μεταρρυθμίσεις που περιμένουν οι πολίτες. Αλλά ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Είδαμε με τη μεταναστευτική κρίση για το ευρώ ότι κολλάμε όταν εφαρμόζουμε με ημίμετρα την ένταξη. Θα πρέπει τώρα να παρουσιάσουμε έργο, να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους μηχανισμούς και τα εργαλεία για να προσαρμοστεί στις προκλήσεις των καιρών. Οπότε ας μην αφήσουμε τους λαϊκιστέ και τους ευρωσκεπτικιστές να μονοπολούν τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα είμαστε, πρέπει να είμαστε ισχυροί, ενωμένοι και να κάνουμε ακόμη ένα βήμα προ μια ευρωπαϊκή φεντεραλιστική δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος Τζάνι για την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι και το Κοινοβούλιο από την αρχή της θητείας αλλά και η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, βασίστηκαν πολύ στην, ε, διάσκεψη, στην οργάνωση αυτής της ε, διάσκεψης ε, λέγοντάς μας ότι αυτό θα αποτελέσει πυλώνα του πενταετούς προγράμματος καθώς επίσης και πυλώνα της νέας θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα από τους ε, εκπροσώπους όλων των ομάδων που αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα αυτής της διάσκεψης. Εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε επιπλέον απαντήσεις ε, γιατί οι πολίτες ε, δεν μας ζήτησαν τον Μάιο μέσω των εκλογών να διοργανώσουμε διασκέψεις, συζητήσεις, φόρα κλπ. Ζήτησαν συγκεκριμένες αποφάσεις, ζήτησαν συγκεκριμένα μέτρα. Άρα δεν τίθεται εδώ ζήτημα να ακούσουμε τους πολίτες. Τους πολίτες τους ακούσαμε. Το πρόβλημα, το πολιτικό πρόβλημα είναι ότι τα θεσμικά όργανα δεν ε, μπόρεσαν, δεν κατάφεραν τα τελευταία χρόνια να δώσουν απαντήσεις ε, στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ε, προβλήματα που σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια, την οικονομική κρίση, τη μετανάστευση. Γιατί αυτό άλλωστε λείπει από, την, από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μπορεί να αγνοηθεί. Πιστεύω ότι τέτοιου είδους ασκήσεις ε, θα μπορούσαν να έχουν έννοια εάν πριν ε, ε, γίνουν προτάσεις αυτό το σώμα μπορούσε να κάνει την αυτοκριτική του σχετικά με τα σφάλματα, τα σοβαρά σφάλματα τα οποία έγιναν στο παρελθόν και που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πλέον μηδενική αξία στη διεθνή σκακέρα. Εάν δεν κατανοήσουμε ότι η πολιτική των τελευταίων 20 ετών στην ουσία μόνο εξασθένησε τα κράτη, μόνο αποδυνάμωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο ε, έφερε περισσότερη φτώχεια στους πολίτες, ε, τότε θα κάνουμε απλώς ε, μία συζήτηση marketing χωρίς καμία έννοια. Ε, πρέπει να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε ε, πού έγιναν τα λάθη. Αλλά μέχρι αυτή την ώρα τα θεσμικά όργανα δεν έκαναν καμία τέτοια προσπάθεια. Ε, αντί να καταλάβουν τα προβλήματα, κάθονται και συζητούν, όπως έλεγε ο συνάλφος των Πρασίνων προηγουμένως, για το φεντεραλισμό ή όχι, για την περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια συζήτηση από τις ταυτότητές ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από την θέση ότι χωρίς τα κράτη μας, χωρίς τους λαούς μας δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος Λεγκούτκο από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για το ψήφισμα, το οποίο θα κληθούμε να εγκρίνουμε από πλευρά του Κοινοβουλίου. Και αυτό που θέλω να πω βασικά είναι το εξή, ότι όλο αυτό το ψήφισμα είναι λάθο. Είναι λάθο. Είναι λάθο, λέω. Γιατί το άρθρο 48, παράγραφος 4 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δηλώνει ξεκάθαρα ότι το Συμβούλιο είναι εκείνο, όχι το Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορούν να συγκαλέσουν τέτοια διάσκεψη, παρά το γεγονός ότι η στάση ε, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ήταν ε, σαφής. Αλλά να θυμόμαστε ότι αποκλίνουμε τελικά από αυτό που ορίζουν οι συνθήκες. Η στάση λοιπόν είναι ότι ο σκοπός ε, αγιάζει τα μέσα. Αλλά να θυμόμαστε ότι αυτό δεν ε, είναι αυτό που ορίζουν οι συνθήκη. Και η διαδικασία παραγωγής αυτού του εγγράφου ήταν επίσης ένα απόλυτο όνειρο. Η συμμετοχή τη Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων, η κατάλογος της ψηφοφορία από πριν, πέντε ομάδες που ψήφισαν αυτό το έγγραφο μυστικά και εξαίρεσαν τις υπόλοιπες ομάδες και την Επιτροπή ΕΜΚΟ. Αν δεν το γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για τυραννία της πλειοψηφίας και για βρώμικο παιχνίδι. Είναι πολύ απλά λάθος. Λάθος γιατί δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον ηγετικό ρόλο στην διαδικασία αυτή προς ζημία των Εθνικών Κοινοβουλίων και η εθνική επικυριαρχία και τα δικαιώματα των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι λάθος επίσης, γιατί δίνει άμα ουσιαστικά την εξουσία σε εκπροσώπους μόνο των πέντε μεγάλων ομάδων. Είναι τυραννή της πλειοψηφίας, ε, γιατί έχει ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα ουσιαστικά. Όπως και σήμερα το πρωί, η διάσκεψη αυτή είναι πολύ απλά ε, το επόμενο βήμα για το επόμενο βήμα στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση σε ό,τι αφορά τους τα ψηφοδέλτια τα υπερεθνικά, το σπίτι στην μεγαλύτερε αρμοδιότητε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εις βάρος των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μην μιλάτε λοιπόν για διαβουλεύσεις, γιατί θα είναι μόνο κατόνομα διαβουλεύσεις. Ο σκοπός είναι ήδη προκαθορισμένος. Και δεν χρειάζεται και τη τρέξη πνάδα για να ε, εξαγάγουμε ότι όλα αυτά θα οξύνουν περαιτέρω τις αποκλήσεις στην Ευρώπη που ήδη είναι ενσυχητικά μεγάλες, αλλά Πάντα ήταν καλή αυτή η υπέρμαχη της ε, ενοποιημένης Ευρώπης για να τα πιέζουν τους άλλους και θα πρέπει να πούμε ότι κανονικά θα πρέπει να νοιαζόμαστε για όλα αυτά, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πιο πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν νοιάζονται. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο Σομπρί, εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ και παραπάνω από ένα μήνα ε, οι Γάλλοι έχουν ε, κατεβεί στους δρόμους και διαμαρτύρονται για την ε, μεταρρύθμιση των συντάξεων και του συνταξιδοτικού Επίσης απεργούν οι γιατροί στα νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οι άνθρωποι όλο και περισσότερο δεν δέχονται μια Ευρώπη χωρίς αλληλεγγύη όπου ε, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον ε, άλλον. Δυστυχώς εδώ μας προτείνεται μια πετσοκομμένη διαδικασία και όσον αφορά τους στόχους και όσον αφορά τη διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ένα πασάλιμα που θα ομορφύνει λίγο την πρόσωψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να, να ε, τολμήσουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους ε, και να αλλάξουμε σε βάθος. Άλλωστε, γιατί δεν αναφερόμαστε στη διάσκεψη αυτή, όχι για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για τη μεταρρύθμιση ε, των ε, συνθήκων. Έχουμε επίσης ε, και ένα μια νέα πράσινη συμφωνία, η οποία δεν μας καλύπτει. Θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη και όχι εμπόριο και ανταγωνιστικότητα. Θέλουμε πραγματική αλληλεγγύη και όχι γενικευμένο dumping. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να παράγουμε δίθεν δημοκρατικές διαδικασίες ε, μέσα από ένα κοινοβούλιο το οποίο και μέσα από μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει πλέον τη λαϊκή νομιμοποίηση για να το κάνει. Ε, δεν πιστεύουμε ότι ε, ε, διασφαλίζεται με τα προτινόμενα ε, η πραγματική ουσιαστική εκπροσώπηση των πολιτών. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν άλλες διαδικασίες μέσω δημοψηφισμάτων κλπ. Δεν είναι δυνατόν να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος της διασκέψεως του 2002 που κατέληξε στην Λισαβόνα. Αντίθετα όμως από τις σαφώς φρασμένες μέσω δημοψηφισμάτων απόψει ε, των πολιτών της Ευρώπης. Βλέπουμε μεγάλη καχυποψία από πλευρά των πολιτών προς ε, ε, τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε θάρρος και να αλλάξουμε τις συνθήκες γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να κυλοπονέσει το βουνό και να γεννήσει ποντίκι. Δεν είναι δυνατόν να μην προχωρήσουμε με ριζικές αλλαγές οι οποίες θα βασίζονται σε σε πραγματικές συμπεριληπτικές διαδικασίες. Θα πρέπει να δώσουμε ουσία στο αρχικό ιδεώδες του αρχικού ευρωπαϊκού οράματος. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των μη ο κύριος Καστάλντο, παρακαλώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, φέτος ε, επιτέλους θα έχουμε την δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης ε, που ως πολιτική δύναμη με επιμονή είχαμε ζητήσει τα τελευταία χρόνια. Ε, βρισκόμαστε ενώπιον του Brexit και νομίζω ότι θα πρέπει να δραχθούμε αυτή τη ευκαιρία έτσι ώστε να οθήσουμε όσο γίνεται πιο ε, φιλόδοξες ε, ε, μεταρρυθμίσεις και να δούμε με μεγαλύτερη αλληλεγγύη το θέμα της μετανάστευσης. Δεν είναι δυνατόν όμως να καταλήξουμε σε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Η διάσκεψη αυτή δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε, ενδεχομένως να οδηγήσει και σε μεταρρύθμιση των συνθήκων μετά από τη διαδικασία ίδιας πρωτοβουλίας που έχει το Κοινοβούλιο. Οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται σε πρώτη γραμμή. Εμεί δε θα πρέπει να είμαστε σαν εκπρόσωποι τους επίσης στην πρώτη γραμμή ε, ε, έκφρασης ε, των προσδοκιών τους και των ελπίδων τους. Δεν πρέπει αυτή η διάσκεψη να είναι απλώς μια επικοινωνιακή διάσκεψη. Για πολλά χρόνια είχε ανεπίτρεπτη αδράνεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες μα αυτή τη στιγμή φοβούνται αλλά και ελπίζουν και μπορούμε να καλύψουμε τι ελπίδε μας μόνο εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τους εκπροσώπους των ε, διαφόρων πολιτικών ομάδων. Βεβαίως, ε, εφ' μπορεί να χρησιμοποιείτε και την μπλε κάρτα. Ε, κύριε Ράνζελ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Συμβούλιο και η Επίτροπος θα ήθελα να πω ότι δέκα χρόνια μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπει στην επόμενη δεκαετία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε βαθύτατες και ευρύτατες εκτενέστατες συζητήσεις για να προετοιμάσουμε τα θεσμικά μας όργανα και γενικώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτό, ε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οργανώνουμε τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι ότι αυτή τη φορά θέλουμε στην προετοιμασία να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να εμπλέξουμε και τους πολίτες σε αυτή τη συζήτηση. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό είναι αυτό που αποκαλούμε συμμετοχική δημοκρατία, όντως. Αλλά προσοχή, δεν θέλουμε να μπερδέψουμε την συμμετοχική δημοκρατία με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Γιατί άλλο είναι να αφογκραζόμαστε του πολίτε, να διαβουλευόμαστε μαζί τους, να τους εμπλέκουμε, να λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη τους στη συζήτηση και άλλο είναι η θεσμική εκπροσώπηση με όλη την παρακαταθήκη που έχουμε από το κράτος δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να διαχωρίζουμε τις δύο έννοιες σαφέστατα. Ακόμη και θα ξεκινήσω ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία με έναν τρόπο που θα χρησιμοποιεί όλη την όθηση και τη συνεισφορά των πολιτών. Πιστεύω ότι και ελπίζω ότι για πρώτη φορά μπορεί να έχουμε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα γίνει ακουστή η φωνή των πολιτών και όπου η γνώμη τους θα μετράει, θα έχει κάποιο βάρος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βίσοφ, για δυόμιση λεπτά. Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίστηκαν από διάφορες συζητήσει ε, κρίσεων, από το Brexit, από πιο μεγάλες και πιο έντονες φωνές των ευρωσκεπτικιστών και των ακρολαϊκιστών. Όχι μόνο εδώ. Η μεγάλη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ το Μάιο πέρσι ήταν ένα πρώτο βήμα για να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Οι πολίτες με την μεγάλη προσέλευσή τους στις κάλπες ξεκαθάρισαν ότι τους ενδιαφέρει η Ευρώπη ότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι για το οποίο διαφορούν, αλλά χρειάζονται και μια Ευρώπη η οποία θα είναι σε θέση να δρά. Δεν είναι κάτι αυτόματο αυτή η συμμετοχή στις εκλογές. Ήταν το γεγονός ότι πολλές ενώσεις ε, ενεργών πολιτών φρόντισαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά από τις άλλες ευρωεκλογέ. Οι πολίτες λοιπόν χρειάζονται μια Ευρώπη η οποία μπορεί να ενεργήσει, μπορεί να δράσει, μπορεί να τους προ... υπερασπιστεί και να τους ενισχύσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό με τη διάσκεψη αυτή επιτέλους να στρέψουμε το βλέμμα προς τα μπροστά και να κάνουμε μια τομή. Αλλά αυτό θα πετύχει μόνο αν τα κάνουμε σωστά, σωστά και τολμηρά θα ήθελα να πω. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η διάσκεψη δεν μπορεί να είναι κάτι, ένα θέμα ρουτίνας. Θα πρέπει να επιτύξουμε το θάρρος και την τόλμη να βγούμε πέρα από αυτά τα οποία μας βολεύουν, να δούμε πού βρίσκεται ο άνθρωπος και αυτός ο πολίτης που αισθάνεται ότι τον έχουμε εγκαταλείψει και να κοιτάξουμε και στην Ήπετρο, να κοιτάξουμε τι πιστεύουν οι ε, εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι εκείνοι που επικρίνουν την Ευρώπη, εκείνοι για τους οποίους η Ευρώπη δεν είναι απαραίτητα σημαντικό έργο. Γι' αυτό είναι σημαντικό λοιπόν οι πολίτες να έχουν άμεση επιρροή από την αρχή και όχι στο τέλος της διαδικασίας να πούνε ένα ναι ή ένα όχι όταν όλα θα έχουν προκαθοριστεί. Γι' αυτό λοιπόν ξεκαθαρίσαμε ότι αυτή η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θεωρούμε ότι αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε μια θεσμική εκπροσώπηση όπου θα συμμετέχουν και πολίτες της ε, Ευρώπης μέσω της Ευρωπαϊκής ε, Οικονομικής ε, και Κοινωνικής Επιτροπής, μέσω της Επιτροπής των Περιφερειών. Χρειαζόμαστε λοιπόν τους δημάρχους, χρειαζόμαστε τους εκπροσώπους του των πολιτών για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω και ζητώ να έχουμε το θάρρος, την τόλμη, να βγούμε από την πεπατημένη και μαζί να διαμορφώσουμε την Ευρώπη με πιο δημοκρατικό τρόπο για να έχει πιο πολλά δυνατότητες δράσεις. Ευχαριστώ, λέει ο Ο κύριος για τρία λεπτά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια και μετά την έναρξη της συντακτικής συνέλευσης και τα τρία θεσμικά όργανα ξανασυμφωνούν για την ανάγκη μιας ε, ρηξικέλευθης μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γεγονός, αυτή η συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων, γιατί έχουν περάσει 20 χρόνια από την έναρξη της προηγούμενης συνέλευσης. Και για πρώτη φορά αυτά τα τρία θεσμικά όργανα λένε όντως είναι απολύτως απαραίτητο να ε, μεταρρυθμίσουμε εις βάθος την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση με τον κύριο Λεγκούτκο, άλλωστε έφυγε στο μεταξύ. Δεν πρόκειται να συζητήσουμε εδώ με τον κύριο Λεγκούτκο. Ο λόγος που έχουμε την διάσκεψη είναι ότι αναγνωρίζουμε ακριβώ τα προβλήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έχουμε το Brexit, μια μεγάλη χώρα που αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δύσκολο κανεί να πει «Α, τέλεια, μια χαρά τα πάμε». Όχι. Υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα όταν μια μεγάλη χώρα εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πέντε χρόνια μετά την έναρξη τη μεταναστευ... Ε, μεταναστευτικής κρίσης δεν έχουμε μεταρρυθμίσει ακόμη το Δουβλίνο. Έχουμε όντω πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν Δέκα χρόνια μετά την ε, χρηματοπιστωτική κρίση δεν έχουμε καταλήξει τραπεζική ένωση, έχουμε πρόβλημα. Και όταν οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί αποφασίζουν τα πάντα στη γειτονία μας, στη Συρία και στη Λιβύη και στην Ουκρανία, τότε έχουμε πρόβλημα. Η πραγματικότητα είναι ότι στο διεθνές προσκήνιο μας χλεβάζει ο Πούτιν, μας εκβιάζει ο Ερντογάν, μας παρενοχλεί ε, ο Τραμπ και η Κινέζικη κυβέρνηση επίσης κάνει τα δικά της. Οπότε ε, ο κόσμος αλλάζει. Ο κόσμος του μέλλοντος θα κυριαρχηθεί από αυτοκρατορίες όπως η Κίνα, η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εμεί δεν θέλουμε να γίνουμε αυτοκρατορία, αλλά θέλουμε να προασπίσουμε μια Ευρώπη όπου όλοι και τα παιδιά μα και τα εγγόνια μα θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτό το νέο κόσμο που θα έχει αλλάξει ριζικά. Και αυτό δεν ισχύει σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε και μέθοδο. Όχι όπως την συντακτική συνέλευση, γιατί η συνέλευση γινόταν με μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, με τον Ζεσκάρ Ντεστέν στην κορυφή, που ήταν πολύ εντυπωσιακό πρόεδρος. Εμείς αυτή τη φορά το αντίθετο πρέπει να κάνουμε. Όχι άνωθεν, αλλά κάτωθεν. Έτσι πρέπει να ξεκινήσει η δική μας διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Από τους πολίτες προς τα πάνω. Και μετά τη γενιά ε, του Μονέτ και του Σούμαν και τη γενιά του Κόλ και του Μιτεράν χρειαζόμαστε μία τρίτη προσέγγιση με το όραμα της πρώτης γενιάς και το θάρρος της δεύτερης γενιάς. Αυτά, ευχαριστώ. Κύριε Βερχόφστατ, δύο συνάδελφοι ζητούν το λόγο για να σας υποβάλουν ερώτηση με τη διαδικασία της γαλάζιας κάρτας, μπλε κάρτας. Δέχεστε ο κύριος Ρόλαντ. Είστε τυχερός σήμερα. Όντως. Νιώθω τυχερός με εσά, κυρία Πρόεδρε, στην έδρα. Ευχαριστώ. Κύριε Βερχόφστατ, μιλήσατε για το μέλλον της Ευρώπης και δική μου βασική ανησυχία για την Ευρώπη και το μέλλον σας είναι η εξάρτηση σε γεωπολιτικό επίπεδο. Αναφέρατε τη Ρωσία του Πούτιν. Ε, πρόσφατα, ο αγωγός ε, Nord Stream 2 που θα φέρει ε, αέριο από την ε, Ρωσία προς ε, τη Γερμανία θα ολοκληρωθεί και μάλιστα και η Δανία έχει υπογράψει. Πώς ε, θέλετε να ανεξαρτοποιηθείτε από τη στιγμή που θα είστε εξαρτημένοι για φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Κύριε Φερχόφστατ, είπατε ότι θέλετε μία προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Παρ' όλα αυτά, αφημολογείτε ότι κάποια κόμματα ήδη έχουν συμφωνήσει για το ποιος θα ηγηθεί της διάσκεψης. Αναφέρεται μάλιστα και το δικό σας όνομα στις φήμες. Διαψεύδετε αυτές τις φήμες και θεωρείτε ότι η ίδια η διάσκεψη θα πρέπει να εκλέξει τον πρόεδρό της. Καλή ιδέα να έχουμε μια δημοκρατική διαδικασία κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. Μακάρι να ψηφίσουν όλοι, να εμπλέξουμε όλου του πολίτε όπω έγινε σε ευρωεκλογέ. Αυτό είναι το καλύτερο. σω θα μπορούσε ο κύριο ασόλη να οργανώσει αυτή τη διαδικασία. Και ίσω υποβάλλω και τη δική μου υποψηφιότητα. Τώρα στους Βρετανούς φίλους θα ήθελα να πω για το Nord Stream 2. Όντω εύστοχο το σχόλιο σα. αλλά το Nord Stream 2 τι αποδεικνύει. Το Nord Stream είναι απόδειξη απουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ελλείψεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα στην Ευρώπη, γι' αυτό έχουμε Nord Stream 2. Οπότε, αν αυτοί όπω και τα μέλη του κόμματο Brexit ε, είναι κατά το Nord Stream, γιατί δεν δημιουργούμε την ε, Ενεργειακή Ένωση, την ε, Ενεργειακή Κοινότητα το συντομότερο δυνατό. Αυτό θα ήταν λύση και το αντίβαρο του Nord Stream 2. Ο κύριο Άλλαρτ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω όχι μονάχα για τα προβλήματα, αλλά για τις ευκαιρίες και τις λύσεις που θα μπορούσαμε να βρούμε στο μέλλον. Αυτή η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ε, έρχεται έγκαιρα ως δημοκρατική διαδικασία τη στιγμή του Brexit ε, έτσι ώστε να προωθήσει την προοδευτική ατζέντα της Ευρώπης. Ε, εμείς ε, θέλουμε να μας δείξουν οι πολίτες εμπιστοσύνη έτσι ώστε να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες ε, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της διάσκεψης. Πρέπει να γίνει η διάσκεψη αυτή γιατί βρισκόμαστε υπό ιστική ε, επίθεση. Η διάσκεψη αυτή είναι ένας τρόπος όλες οι χώρες να προχωρήσουν προς τα εμπρός, ακόμα και τα μελλοντικά, ε, ε, οι χώρες που μελλοντικά θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σκοτία και ελπίζουμε και άλλα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου να ακολουθήσουν και να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αναπτύξει στη Σκοτία ε, μία ε, καινοτόμα ιδέα ότι ε, ασχέτως από πού προέρχεται ο πολίτης, ασχέτως από που ανήκει ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα σε δημοκρατικές διαδικασίες και έχει δικαίωμα ε, σε αλληλεγγύη. Στην ε, Σκοτία βασιζόμαστε στο κράτος δικαίου το οποίο βασίζεται ε, στις ευρωπαϊκές αρχές και επομένως η Σκοτία προσβλέπει να είναι μελλοντικά μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μπέκ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το 2000 ξεκίνησε η διαδικασία της Λισαβόνας ε, έτσι ώστε ε, η Ευρώπη και παραθέτω να γίνει ε, η πιο προωθημένη οικονομία βασισμένη στην γνώση. Όσο πλησιάζαμε στο 2010 άρχιζε η μετονομασία στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Έφτασε όμως και το 2020 ε, και αυτή η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία που θα ήταν ο ηθικός πρωταθλητής ε, του, της, ε, του πλανήτη με το υψηλότερο εισόδημα και την καλύτερη διαδικασία είναι αυτό που έχει την μικρότερη ανάπτυξη και τον με υψηλότερο εταιρικό φόρο και λοιπά. Τα οικονομικά στοιχεία στοιχεία δε ε, επιδεινώνονται ε, και ε, ακόμα περισσότερο και για τις πιο ευάλωτες χώρες και αυτές που δεν ανήκουν στο ευρώ. Τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση για την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης για να κάνουμε πιο δημοκρατική την Ευρώπη. Γίνεται λόγος για την οικονομία αλλά προστίθενται νέοι φόροι και ένα Green Deal που θα κοστίσει πάνω από ένα τρεις και ε, στο όνομα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής ε, ζητούμε όλο και περισσότερους ε, μη Ευρωπαίους να έρθουν στην Ευρώπη έτσι ώστε να γίνει λιγότερο ευρωπαϊκή η Ευρώπη. Ο Σίγμουν Φρόιντ μίλησε για τη διαφυγή μέσω της ε, ασθενείας ε, ε, και, για, και εδώ αντιμετωπίζουμε μια νευρωτική αποφυγή της πραγματικότητας. Ο νευρωτικός ασθενής στην ουσία θέλει να παραμείνει ασθενής. Υπάρχει μήπως καλύτερη διάγνωση για την Ευρώπη, την σημερινή Ευρώπη η οποία ενώ αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα ε, και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην ουσία θέλει να ξεφύγει από την πραγματικότητα παίρνοντας φάρμακα και ναρκωτικές ουσίες ε, που θα τις κοστίσουν ακόμα περισσότερο. Για 1,5 λεπτό, κύριο Κρασνοντέμσκι. Παρακαλώ, όχι σφυρίγματα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι μόνο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη υπήρχε και πριν την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην το ξεχνάτε και κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει Ευρώπη ακόμη και αν διασπαστεί, εξαφανιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα, δημιουργηθούν άλλες μορφές διεθνούς συνεργασίας. Οπότε θα πρέπει έχοντας υπόψη αυτή τη διαφορά να σκεφτούμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχουμε πολλούς ε, βαθιστόχαστους ε, διανοούμενους και αριστερούς και δεξιούς που διαπιστώνουν ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός βρίσκεται σε μια κρίσιμη ε, στιγμή. Οπότε είναι λογικό να χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Είμαστε υπέρ μιας ειλικρινούς, έντιμης, ανοιχτής συζήτησης και να μην αναφέρονται τόσο μαυρά άσπρα οι πολέμοι της ευρωπαϊκής ένταξης. Δεν θέλουμε να διχάζουμε για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε καλούς και κακούς ε, Ευρωπαίους. Γιατί μερικοί μίλησαν για φεδεραλιστική δημοκρατία. Στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εμπλέξουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να τους προσετεριστούμε. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή ενιαία δημόσια σφαίρα. Και οι συζητήσεις σίγουρα με τους πολίτες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις ε, συζητήσεις στο ε, Ευρωπαϊκό, στο, στα κοινοβούλια αλλά να έχουν συμβουλευτική ισχύ. Αλλά ας μην ξεχνούμε το άρθρο 48 Τη ε, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριο Κύριε Σόλτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αφήνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τον ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ε, διαδικασία αυτή που θα πάρει περίπου δύο χρόνια. Αυτό είναι θετικό και με το σημερινό ψήφισμα το Κοινοβούλιο προβάλλει το θέμα αυτό στην ευρωπαϊκή δημόσια γνώμη σε ό,τι αφορά τους στόχους, τη μορφή και τις μεθόδους για το πώς θα γίνει η συνεργασία με τους Ευρωπαίους πολίτες για μια νέα καθορισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων του μέλλοντος και των καθημερινών προβλημάτων μετά από χρόνια υπόδεινων κρίσεων. Θέλουμε να αποφασίσουμε από κοινού ποια Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε και θέλουμε και πώς θα πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και πιστεύω ότι είναι πολύ βασικός αυτός ο στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να δώσουμε στους πολίτες την ε, κεντρική, τον κεντρικό ρόλο για να υπάρξει η συμμετοχική δημοκρατία και η συμμετοχή των πολιτών για την επιτυχία της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής και για ενεργή διάλογο και μια στενή συνεργασία. Και μια διάσκεψη για τη μέρα της Ευρώπης καταρχάς σημαίνει ότι θα πρέπει στους πολίτες να δώσουμε απάντηση στις προσδοκίες τους και στα νερά τους. Αυτοί θα πρέπει να αποφασίσουν ποια θέματα θα πρέπει να πραγματευτούμε προκειμένου να κλείσουμε τα δημοκρατικά ελλείμματα, να καταρτήσουμε νέες πολιτικές στρατηγικές και να βελτίσουμε την καθημερινότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εθνικό επίπεδο και σε αυτούς τους εκπροσώπους του ID και του ECR. Γιατί φοβόσαστε τους πολίτες αυτούς οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν και να προωθήσουν ευρωπαϊκό έργο στην ε, Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν διαφάνεια και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η διάσκεψη και η συζήτηση να ξεπεράσει τη διάσκεψη. Κύριε Παπαδάκη, για ένα λεπτό. αλήθεια από πού και ως πού μιλάτε για το μέλλον της ευρώπης ταυτίζοντάς το με το μέλλον της ευρωπαϊκής ένωσης μιας ένωσης των μονοπωλίων που κάποιοι πρόβαλαν κάποτε ως αιώνια ως νομοτέλεια και σήμερα καταγράφονται brexit φυγόκεντρες τάσεις αντιθέσεις ενώ στα ίδια τα κείμενά σας ανησυχείτε για την ανεμική καπιταλιστική ανάκαμψη. μεθοδεύεται μια χρυσοπληρωμένη εκστρατεία πλήση εγκεφάλου προκλητικού εξοραϊσμού της ευρωπαϊκής ένωσης χειραγώγησης και αντικομουνισμού επιχειρώντας να αναχαιτίσετε την εντυνόμενη αμφισβήτηση και έλλειψη εμπιστοσύνης των λαών και της νεολαίας αυτής. αυτήν. στείνονται διασκέψεις δήθεν λαϊκής συμμετοχής με επιχειρηματικούς ομίλους μικιό λόμπι και εργατοπατέρες αντίθετα από ό,τι ισχυρίζεται και η γκουε που συνυπογράφει το σχετικό ψήφισμα ως γνήσιος απολογητής της η ευρωπαϊκή ένωση δεν αλλάζει ούτε όπως ισχυρίζονται οι ακροδεξιοί κάνει λάθη υπηρετεί ανεπίστρεπτα το εκμεταλλευτικό σύστημα είναι αντίπαλο των εργατικών λαϊκών συμφερόντων διαρκή υπονομευτή της υπεράσπισης συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων. το δικό τους μέλλον μπορούν να χαράξουν οι λαοί με αποδέσμευση από την ευρωπαϊκή ένωση με το λαό στην εξουσία για την ευρώπη του σοσιαλισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ε, κάτι τυχαίο, αλλά ένα ειρηνευτικό όραμα κατά των ε, φρικαλαιοτήτων του πολέμου. Είμαστε ε, η πρώτη γενιά που δεν βίωσε πόλεμο, αλλά δεν ξέχασε τον πόλεμο. Είναι μια ειρηνευτική διαδικασία, ένα σχέδιο ειρήνης Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάποια στιγμή σταμάτησε και άρχισε να παρεδρομεί. Στο παρελθόν ήταν ένα όνειρο, αλλά σήμερα είναι μια πραγματικότητα που δεν ικανοποιεί. Θα πρέπει να ζούμε το όνειρο, αλλά Ζούμε καιρούς που οι πολιτικοί δεν έχουν νομιμοποίηση για να ονειρεύονται και μερικές φορές ε, γίνονται γνωστοί ως ε, ε, φλίαροι με κενά λόγια και σλόγγαν. Θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε κοντά στους πολίτες και αυτοί μας εξέλεξαν και στις προεκλογικές εκστρατείες όταν μιλούμε με τους πολίτες και όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε πολίτες οι ε, αν δεν εκπροσωπούμε του πολίτε, τι κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και οι συνελεύσει των πολιτών, παράλληλε ε, με τα κοινοβούλια, ουσιαστικά δίνουν ομοιοποίηση στα κοινοβούλια η Ευρώπη δεν χρειάζεται πολιτικούς που ονειρεύονται θεροβάμονες. Θέλουν πολιτικούς που πιστεύουν, που πιστεύουν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς εθνικισμούς, χωρίς σύνορα, χωρίς διακρίσεις, που πιστεύουν ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που πιστεύουν ότι μαζί θα γίνουμε καλύτεροι, που πιστεύουν σε μια φεντεραλιστική Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν ποια θα είναι η πορεία μας, προς τα που οδεύουμε. Ε, σε τι Ευρώπη πιστεύουμε θα πρέπει να αποφασίσουμε και όχι τι Ευρώπη ονειρευόμαστε. Ευχαριστώ. Κύριε Γκονσάλες Πόνς, κάποιος συνάδελφος ε, ζητά με τη διαδικασία της μπλε κάρτας ε,